και θα χορηγήσω, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν σήμερα στους αρμόδιους. Είναι η τελευταία ολομέλεια του έτους και χαίρομαι που εργαστήκαμε επικοδομητικά και αυτή τη φορά σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και ελπίζω να μπορέσω